Καλημέρα σας. Νομίζω πως τώρα λειτουργούν όλα με τη διερμηνία. Εάν λοιπόν όλα λειτουργούν σωστά, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας. Έχετε όλη την ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχουν τροποποίησει. εγκρίνεται λοιπόν. ανακοινώσει τη Προέδρου, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο και περνάμε στην ψηφοφορία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την γνωμοδότηση του κυρίου Σάβαρμα για την πορεία της συζήτηση ε, για το μέλλον της Ευρώπης. Θα θέλατε το λόγο? Θέλετε το λόγο, κύριε Σιγητά? Όχι. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες ψηφοφορίας και ξεκινάμε με το μέλλον της Ευρώπης. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά ο, αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα την τροπολογία 21. 21. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Α, κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 25. Πέρας. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο, πολύ ωραία. Ελέγχουμε την 29. Πέρας, απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ. Με προφορική τροπολογία δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 35 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα. Τρία τμήματα, με συγχωρείτε, λέει πρόεδρο. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά θα το δούμε, δεν ήταν σαφές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39. Με προφορική τροπολογία δεν υπάρχουν ενστάσεις υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40. Υπέρ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 κατά. 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την τροπολογία 3. Απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφοφορία με ονομαστική κλίση για το ψήφισμα που έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 19 ψήφους υπέρ, μία κατά. Συγχαρητήρια. Σχέδιο γνωμοδότηση στην Επιτροπή Ήτρε. Κυρία Λαμπαγιώβα, η Ε, θέλετε το λόγο? Όχι. Περνάμε λοιπόν αμέσω στην ψηφοφορία. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές μπορούμε να ελέγξουμε. Τροπολογία 30. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33. Ναι, θέλετε έλεγχος 32. Τέλος, εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 4. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Η 4 εγκρίθηκε. Να ελέγξουμε. Για την 4 ψηφίζουμε. Ναι, εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8 και 36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 Περά εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και ψηφίζουμε με νομιστική ψηφοφορία το σύνολο της γνωμοδότησης άρχεται ψηφοφορία και εγκρίνεται 22 υπέρ 0 κατά. Συγχαρητήρια στην συγγήτρια. Περνάμε τώρα στην ε, ονομαδότηση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Ο κύριο Πυρίνσκι είναι ο εισηγητή. Α, συγγνώμη. Έχουμε δύο φακέλους στη ΣΥΤΡΕ. Η κυρία Τλαπαγιώβα η συγγήτρια δεν θέλει το λόγο. Περνάμε στην ψηφοφορία για το πρόγραμμα πλαίσιο έρευνες και κοινοτομίες. και ξεκινάμε με την τροπολογία 11. Ξέρετε όλοι που είμαστε. Υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε. Πέρα συγκρίνεται. 12. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Uh, amendment 1. Ένα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 14, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται... 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 με τεχνική τροπολογία υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται... 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές, λογικά απορρίπτεται να ελέγξουμε, γιατί δεν είμαι σίγουρη. Λήξη, εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ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 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ίσως, αλλά να ελέγξουμε. 28. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 32. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 41 καταπίπτει. Να ελέγξουμε τη 42. Για να ελέγξουμε τη 42 παρακαλώ. Ελέγχουμε την 42. Ποιος λείπει. Τέλος. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 41, 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Μάλιστα. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 52. Τέλος. Λυπάμαι. Ίσως ήταν πολύ γρήγορο. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 53. Εγκρίνεται. Λυπάμαι. σχόλιο εκτός μικροφώνου και απαντάει η για να, τα, για να είμαι ειλικρινή, το ίδιο σκέφτηκα. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Να ελέγξουμε την 54. Απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στη λογική σκέψη 9, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται και 7, υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται και άρχεται η ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου, ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται με βρία πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Τώρα περνάμε στο σχέδιο γνωμοδότησης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Ο κύριος Πυρίνσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείναμε μία απεριεκτική αναθεώρηση αυτού το οποίο προτείνει η Επιτροπή και συνειδητοποιώ ότι λόγω έλλειψης χρόνου και ευκαιρίες να εξηγηθεί με, περισσότερες λεπτομέρειες ενδεχομένως υπάρχουν κάποια ερωτήματα και έλλειψη σαφήνες. Ε, όπως παρατηρήσατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, να παρουσιάσαμε την έκθεση αυτή, πράγματι είναι μια περικτική παρουσίαση αυτό το οποίο προτείνει η Επιτροπή. Ενδεχομένως υπάρχουν δισταγμοί προκειμένου να υποστηριχθεί το σύνολο του κειμένου και βεβαίως αυτό θα φανεί και στην ε, ψηφοφορία αλλά θα πρότεινα να εγκριθεί η γνωμοδότηση και να, αποσταλ... πάει στην έμπλε. Γιατί μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πραγματικά περιλαμβάνει πολύ σκληρή εργασία και επαλήθευση και ε, διασταύρωση ε, των άλλων νομοθετημάτων, ε, σχεδίων νομοθετημάτων τα οποία θα ψηφιστούν την προσεχή περίοδο και θεωρώ ότι είναι αναγκαίο για τις προτάσεις και τις γνωμοδοτήσεις μας να μην ε, χαθούν. Γι' αυτό πραγματικά θα το εκτιμούσα αν το στηρίζατε στο σύνολό του. Ευχαριστώ πολύ. Η 104 έχει αποσύρθει η τροπολογία περθών 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Επαλήθευση για την 6 παρακαλώ. Λείπει μία ψήφος. Πέρας του ελέγχου. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, Επαλήθευση παρακαλώ για την ένα. Απορρίπτεται. Εκτός μικροφώνου. Ο μιλητής είναι εκτός μικροφώνου. Πρόεδρος, υπήρξε μια πλατιά πλειοψηφία υπέρ για την 5. Συμβαστική 1 απορρίπτεται. 7. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ για την 7. Απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση παρακαλώ για την 105 Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Θα το ελέγξω. 2 παρακαλώ. Συμβαστική 2. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές Τη 10 παρακαλώ, επαλήθευση. Απορρίπτεται. Η 11 καταπίπτει. 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική υπαριθμών 3. Επαλήθευση. Ίσως έτσι μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρόνο. Για την τρία λείπει μια ψήφος. Εγκρίνεται λοιπόν 106 υπέρ. 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 και 11 καταπίπτουν 112 συνεπώς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση παρακαλώ για τη 13 Όλοι θα πρέπει να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 18 έχει αποσυρθεί 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική υπαριθμών 3 α όχι συγγνώμη λέει πρόεδρος 23 δηλαδή καταπίπτει 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ όχι καταπίπτει λυπούμε 117 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 έχει αποσυρθεί. 119 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 η 35 έχει αποσυρθεί 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 122 υπέρ, κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίθηκε έλεγχος 122 εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52, η 52 έχει αποσυρθεί, 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 133 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 57 υπέρ, α, έχει αποσυρθεί 134 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 136 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται ένα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται δύο υπέρ, επαλήθευση για την ένα. Πέρας της επαλήθευσης. Εγκρίνεται, λυπούμε λέει η πρόεδρος, δύο υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 77 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται 3 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται 70 Νομίζω ότι κάποιος, ε, κάποια ψήφος λείπει. Πέρας της επαλήθευσης εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει. 79 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση παρακαλώ για την 80. Πέρας. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές. 82 έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ κατά να γίνει επαλήθευση για την 83. Ωραία, καλώς. 83 έλεγχος. Πέρασε ψηφοφορίες, εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ για την 90 να γίνει παλήθευση. Όχι, για την 89 λέει η πρόεδρος. Έλεγχος. 89. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται λοιπόν. 90 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά... επαλήθευση παρακαλώ για την 91. Απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ. 93 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την 93 εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχ... επαλήθευση για την 97 απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει απορριφθεί να γίνει επαλήθευση παρακαλώ για την 103 Λείπουν δύο ψήφοι, παρακαλώ εγκρίνεται. Το σύνολο της ε, γνωμοδότησης έτσι όπως ε, τροποποιηθεί ε, με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία για την γνωμοδότηση Ναι, με 20 ψήφους υπέρ και μία κατά εγκρίθηκε. Το είδα εδώ, ξέχασα να σας το πω, με συγχωρείτε, λέει ο Πρόεδρος. Περνάμε στην ψηφοφορία για την γνωμοδότηση του Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Ξεκινάμε με την τροπολογία 40. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 41, υπέρ, κατά. Ελέγχουμε τη 41, ηλεκτρονικά. Πώς είπατε? Εκτός μικροφώνου το σχόλιο. 41 λοιπόν. Απορρίπτεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε. Νομίζω πως απορρίπτεται. Σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. Λάθος έκανα. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46. Καταπίπτει. 46. 47. Υπέρ. Κατά. Οι 44 εγκρίθηκαν. Εγκρίθηκε και οι 45 Ας ψηφίσουμε. Τη 46, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Χρειάζεται, να είναι σαφέστερος ο κατάλογος ψηφοφορίας. 47, υπέρ. Κατά. Αποχές, μπορούμε να ελέγξουμε Ελέγχουμε τη 47. And, uh, the check is over. Πέρας. Α, όχι, μας λείπει ένας. Εγκρίθηκε. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λογικά, αλλά ας ελέγξουμε τη 12 ηλεκτρονικά. Μας λείπει μία ψήφος ακόμα. Πέρας. Απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ελέγχουμε την 57. Πέρας. Απορρίπτεται, δεν το είδα. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. 65 έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 66. Πέρας. Όλοι είστε υπέρ. Ωραία. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. 17 ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θα ελέγξουμε την 71 νομίζω πως εγκρίνεται όμως ελέγχουμε την 71 μας λείπουν δύο. εγκρίθηκε 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά αποχές Ας ελέγξουμε και την 77, για να είμαστε σίγουροι. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται και αυτή νομίζω. Θέλετε έλεγχο. Ωραία, ας ελέγξουμε την 78. υπέρ, 79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται, αλλά ελέγχουμε. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Ωραία. Ψηφίζουμε την 26. Μας λείπει μία ψήφος και είναι σημαντική. Όλοι πρέπει να ψηφίσετε. 11, 11 προ 11. 27, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά απόχέ. απορρίπτεται. Πάλι 11 προς 11, αλλά θα ελέγξουμε αν το θέλετε. Αν συμμετάσχετε όλοι, είναι 11 υπέρ, 11 κατά. Αλήθεια. Απορρίπτεται. Το είδα το αποτέλεσμα. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε τη 35. Απορρίπτεται. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά απόχέ. απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 10 υπέρ κατά αποχές... Όχι, θέλω τα ελέγχω. Δεν είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την γνωμοδότηση με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Μας λείπει μία ψήφος, ονομαστική κλίση. Θα πρέπει να είστε και στον κατάλογο της ψηφοφορίας στο τέλος. Μάριαν, ψήφισες. Μας λείπει ένας. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ωραία. Ψήφισαν όλοι 19 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια σχέδιο γνωμοδότησης ε, για το Ίντερεγκ. Ο κύριος ε, Κον είναι ο συγγετής. Θέλετε το λόγο. Όχι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είστε έτοιμοι. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται να ελέγξουμε την 30. Τώρα έχουμε 23. Ποιος ήρθε. Θεέ μου. 22. Mm. Mm. still 22. Εξακολουθούμε να είμαστε 22, κάποιος λείπει. Τέλος της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε τη 33. Πέρας. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά Εποχές. απορρίπτεται. Συγγνώμη, 34. Όχι. 2. Μάλιστα, πρέπει να ελέγξουμε τη 2. Δεν μπορώ να καταλάβω που είναι η πλειοψηφία. Πέρας. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Εποχές να ελέγξουμε. Τριάντα τέσσερα. Πατήστε το κουμπί. Ξεκολουθούν να λείπουν δύο άτομα. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρία υπέρ. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε την 9. Πέρας. Απορρίπτεται. 10 υπέρ 37, συγγνώμη. Υπέρ. Κατά αποχές γκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά αποχές γκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40. Υπέρ κατά εποχές. Λογικά θα πρέπει να εγκρίνεται ή να ελέγξουμε τη 40. Απορρίπτεται. Λυπάμαι. 12 υπέρ. Κατά εποχές. Να ελέγξουμε και τη 12. Ψηφίζουμε για τη 12. Πάλι λείπει μια κάρτα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 κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά να ελέγξουμε την τροπολογία 1 λήξη εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ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 να ελέγξουμε την 27. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Ελέγχουμε την 27 και εγκρίνεται. Και περνάμε στην ψηφοφορία, την ενομαστική για το σύνολο του κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 19 υπέρ, 0 κατά και 2 εποχές. Τώρα Περνάμε στην τελευταία γνωμοδότηση για σήμερα. Γνωμοδότησή μα στη Γιούρη και στη Λίμπε, ο κύριο Ντε Είναι ο εισηγητής Ντένι. θέλει το λόγο? Όχι, να περάσουμε. Στην ε, τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχέ. ακρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε τη 10. Και πάλι κάποιος λείπει. Πιέστε το κουμπί. Εγκρίνεται. 53 καταπίπτει, 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 54 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά εποχές συγκρίνεται, 55 υπέρ κατά εποχές συγκρίνεται 12 υπέρ κατά εποχές συγκρίνεται 13 υπέρ κατά εποχές συγκρίνεται 14 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά εποχές συγκρίνεται 16 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 17 υπέρ η 16 απορρίφθηκε. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 καταπίπτει. 19 σε δύο μέρη. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1. Υπέρ. Για την 1. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε τη 2.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 Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 36. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται 36. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 5. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. 37 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Καταπίπτει. Πάμε 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, 44 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, 45 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται, 46 υπέρ κατά αποχε εγκρίνεται, 7 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 7. Εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ψηφίζουμε το σύνολο της νομοδότησης, με ονομαστική ψηφορία, άρχεται η ψηφοφορία. 20, συγγνώμη, 19 προς 1. Συγχαρητήρια στον εισηγητή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώνουμε εδώ τη συνεδρία. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα στις 3, για την ακρόση της κυρίας Κρέτσου.